δήλωση της Κομισιόν για το θέμα προστασία πληροφοριοδοτών και δημοσιογράφων για φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή για την Κομισιόν. Πρώτη έχει το λόγο η κυρία Γιούροβα για να κάνει μια δήλωση. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης είναι πολύ σημαντικό για τους δημοσιογράφους και όσους εργάζονται στα μέσα ενημέρωσης. Θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να ασκούν κριτική χωρίς να φοβούνται διώξεις. Πρόκειται για ένα βασικό χαρακτηριστικό της δημοκρατικής κοινωνίας. Ίσως είναι δυνατόν να περιοριστεί η ελευθερία έκφρασης, αλλά μια τέτοια προσπάθεια περιορισμού θα πρέπει να είναι αναλογικά τεκμηριωμένη και δεν θα πρέπει ο περιορισμός ε, να ξεπερνά κάποια όρια ανάλογα με τις συνθήκες. Δεν υπάρχει ένα αρμονισμένο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία αυτών που κάνουν καταγγελίες, που προβαίνουν σε καταγγελίες. Αλλά υπάρχει η περιγραφή αυτής της ιδιότητας σε ορισμένους τομείς όπως το δίκαιο του ανταγωνισμού και επίσης ο κανονισμός για καταχρήσει στις αγορές και ιδιαίτερε χρηματαγορές. Αυτοί οι οποίοι ε, παρέχουν πληροφορίες και αναφερόμαστε σε αυτούς που παρέχουν πληροφορίες προς τις δημόσιες αρχές. Θα πρέπει λοιπόν τα ίδια τα κράτη-μέλη να ρυθμίσουν την περίπτωση αυτή σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία στα πλαίσια των κανόνων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ε, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Vielen ευχαριστώ. Περνάμε τώρα σε προσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων για το ΕΛΚ η κυρία Ρωμάνα Τόμς για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνούμε όλοι πως η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, επηρεάζει την οικονομία μας και το επίπεδο ζωής μας. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι το ασφαλές νέφος, ένα μέσο του διαδικτύου, μέσω του οποίου μπορούμε να μοιραστούμε πληροφορίες για αυτές τις πρακτικές. Ακούγεται πολλά υποσχόμενο, όταν όμως φτάνουμε στο θέμα της εφαρμογής υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Ειδικά νομικής φύσης. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Δηλαδή το θέμα της ε, προστασίας ε, προσωπικών ε, δεδομένων. Εν ολίγης, όταν λαμβάνονται αποφάσεις στο μέλλον, θα πρέπει στο Κοινοβούλιο να γνωρίζουμε τον ρόλο μας, ότι είμαστε δηλαδή συνομοθέτες. Και πρέπει να αναρωτηθούμε, θέμε να πάμε πέρα από αυτό το ρόλο ή όχι. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό για τους σοσιαλδημοκράτες Πέτερ Σιμών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, συμφωνούμε με την Κομισιόν. Υπάρχει στο δίκαιο του ανταγωνισμού και αλλού κάποιες ειδικέ διατάξεις. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Πιστεύει κάποιος εδώ πέρα στην αίθουσα πως τα κράτη-μέλη θα τα κάνουν αυτά τα πράγματα από μόνοι τους, δηλαδή θα βρουν το σημείο ισορροπίας μεταξύ του, ε, νομικού, του νόμιμου συμφέροντος των εταιριών περί εμπιστευτικότητας και του ένομου συμφέροντος ε, της κοινωνίας ε, να μάθει για την ε, φοροδιαφυγή Αν τα αφήσουμε στα κράτη-μέλη θα αποτύχουν. Γι' αυτό πρέπει να είστε θαραλέοι. Πρέπει ακριβώς να υπάρξει μια ενιαία ευρωπαϊκή αντίληψη για το πότε μπορεί να γίνει αποκάλυψη τέτοιων μυστικών όταν δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η κοινωνική τους σημασία ώστε υπερισχύει της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας και δεν υπάρχουν κυρώσεις. Τέτοια πρόταση περιμένουμε από σας. Ως ακριβώς ε, θεματοφύλακες των συνθήκων Οφείλεται, δηλαδή να δείτε πως ε, υπάρχει μια συνένεση θεωρώ εγώ στην Ευρώπη για αυτό το θέμα που απαιτεί από την Κομισιόν να ε, καταθέσει τόσο θαραλέες προτάσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους για δύο λεπτά, Μαριαν Χάρκιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ομάδα η οποία θα ξεκινήσει για τα θέματα αυτά αύριο το απόγευμα θα είναι χρήσιμη ελπίζω για να προστατεύσουμε ε, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι προβαίνουν σε καταγγελίες ε, για το κοινό συμφέρον. Η συγκεκριμένη αυτή κατηγορία φυσικά δεν αρκεί για να αποτρέψουμε κάθε μορφή διαφθοράς ε, στη δημόσια διοίκηση. Μέχρι τώρα, στο αίτημα του Ευρωπαίου Ομπουτσμαν, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για να υπάρξουν εσωτερικοί κανόνες σε σχέση με τις καταγγελίες και για την προστασία αυτών που προβαίνουν στις καταγγελίες, από, τα, από τις εννέα κοινοβουλευτικές διοικήσεις, μόνο, ε, μάλλον κοινοτικές διοικήσεις και όργανα, μόνο δύο έχουν ανταποκριθεί με θετικό τρόπο. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή κατάλληλο νομικό πλαίσιο κοινοτικό. Ε, τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα, αλλά τίποτα άλλο δεν μπορεί να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λόγω ακριβώς ε, της ύπαρξης αυτών των ανθρώπων που κατήγγυλαν τα LuxLeaks δημιουργήσαμε την Ειδική Επιτροπή ε, για τις φορολογικές επιμέρους ρυθμίσεις θα πρέπει να κατανοήσουν και οι κυβερνήσεις ότι προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τη δικαιοσύνη και στον τομέα της φορολογίας. Σε όλα τα επίπεδα η διαφθορά δυστυχώς θα περνά απαρατήρητη αν δεν διευκολύνουμε τις καταγγελίες. αν γνωρίζουν αυτοί που μπορούν να καταγγείλουν θα είναι ασφαλείς ή μάλλον δεν γνωρίζουν ότι θα παραμείνουν ασφαλείς, τότε δεν θα ε, δημοσιοποιηθούν οι καταγγελίες ε, και η διαφθορά θα συνεχιστεί. Έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Νεγκρέσκου, θα, θα απαντήσετε. Κύριε Νεγκρέσκου, έχετε το λόγο. Μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από αυτά που είπατε αλλά θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα κάτι για τους φοροφυγάδες. Υπάρχουν φοροφυγάδες οι οποίοι μετά γίνονται πληροφοριοδότες κατά άλλων. Αυτούς ή θα τους κάνουμε. Δεν κατάλαβα καλά νομίζω τι εννοούσατε. Είπατε για φοροφυγάδες οι οποίοι γίνονται πληροφοριοδότες για άλλους. Εγώ αυτό άκουσα. Δεν καταλαβαίνω όμως τι σχέση έχει αυτό το ερώτημα τέλος πάντων. Η φοροδιαφυγή είναι έγκλημα, αδίκημα, έγκλημα και φυσικά πρέπει να υπάρξει τίμημα. Αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτε άλλο γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί το θέσατε αυτό. Αν το καταλάβαινα θα μπορούσα να σας δώσω μια καλύτερη απάντηση. Ίσως να το δούμε αργότερα άλλη φορά. Ευχαριστώ. Για τους ε, φιλελεύθερους, ε, να μισή λεπτό, κύριος ε, Ντεμάζη. Κύριε Πρόεδρε, η Γκουε ζήτησε αυτή την συζήτηση και ευχαριστώ τους συναδέλφους. Ο δημοσιογράφος Εντουάρ Μπερέν κατηγορήθηκε στο Λουξεμβούργο επειδή αποκάλυψε τα όσα περιείχαν οι LuxLeaks που αφορούσαν τις φορολογικές συμφωνίες των αρχών με τις εταιρείε. Δεχόμαστε βεβαίω το δίκαιο του Λουξεμβούργου αλλά και την ελευθερία του τύπου. Εδώ πέρα παραβιάζεται το δικαίωμα της ελεύθερης πληροφόρησης όπως αυτό το ορίζει η ΕΣΔΑ και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν είναι ε, δυνατόν να υπερισχύει εδώ πέρα η εμπιστευτικότητα και τα εμπορικά μυστικά των εταιριών. Χάνεται κάθε χρόνο ένα δισεκατομμύριο σε φορολογικά έσοδα ή, ή φοροδιαφυγή με συγχωρείτε, δεν είναι εμπορικό μυστικό, δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να προστατεύονται νομικά οι πληροφοριοδότες όταν βεβαίως αποκαλύπτουν πράγματα τα οποία είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Η Κομισιόν δε του κυρίου Γιούνκερ είναι υπό την ηγεσία ενός ανθρώπου ο οποίος είναι υπεύθυνο για την νομοθεσία αυτή στο Λουξεμβούργο. Αναμένω λοιπόν επιτέλους να υποβάλει τις σωστές προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου όπως κάνει και οι άλλες περιοχές του κόσμου και να μην προστατεύει τους εγκληματίες. Σας ευχαριστώ και για το ότι μείνατε εντός του χρόνου η πράσινη. Τώρα η κυρία Ζολή για ένα λεπτό. <clears throat> Κύριε Πρόεδρε, στις 23 Απριλίου ο Εντουάρντ Περέν, δημοσιογράφος που είχε αποκαλύψει το σκάνδαλο, ε, μεγάλο τμήμα του σκάνδαλου LuxLeaks, διώχθηκε από την Λουξεμβουργική Δικαιοσύνη. Ο Αντουάν Τελτούρ για παραβίαση του επαγγελματικού μυστικού. Αυτά είναι επιθέσεις κατά της δημοκρατικής ζωής. Ως προς την φορολογική δικαιοσύνη αλλά και τα εργασιακά, ο ρόλος των πληροφοριοδοτών και των ε, δημοσιογράφων είναι ζωτικός. Ενώ ακούγονται τόσα πολλά για διαφάνεια λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία της για το επαγγελματικό μυστικό επέλεξε να μην υπάρξει διαφάνεια. Κυρία Επίτροπε, η περίπτωση του Εντουάρ Περέν και του Εντουάρ Ντελτούρ είναι απαράδεκτες διώξεις. Θα έπρεπε να θεωρηθούν ήρωες και να προστατευθούν ενώ θέλετε και στα 28 κράτη-μέλη να εφαρμοστούν απαρχαιωμένοι νόμοι για να προωθήσετε τα συμφέροντα ορισμένων εναντίον του γενικού συμφέροντος. Γνωρίζουμε τα ονόματα που έχουν αυτά τα ιδιωτικά συμφέροντα. Γνωρίζουμε τους λομπιίστες και η καινούργια επιτροπή και η καινούργια επίτροπος θα ήταν προς τιμήν να ρίξουν άπλετο φως σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρόεδρε, σήμερα στο Κοινοβούλιο συζητάμε την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Δημιουργήσαμε και μία ειδική επιτροπή γι' αυτό. Όλα αυτά κατέστησαν εφικτά χάρη στην παρέμβαση δημοσιογράφων και πληροφοριοδοτών όπως τον Αντουαντελτούρ. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να προστατεύουμε αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν να δημοσιοποιούν απαράδεκτες και στρεβλές καταστάσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των φορολογικών. Όταν κάποιος θέλει να εμβαθύνει τέτοιου είδους έρευνες και θέλει να δημοσιοποιήσει στοιχεία τα οποία έχει στην κατοχή του, πρέπει να έχει και τις εγγυήσεις να το κάνει χωρίς συνέπειες. Είναι αλήθεια ότι πολλοί από τους πληροφοριοδότες αυτούς ήταν συνένοχοι κάποιων πρακτικών παρανόμων. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει πράξεις πολύ πιο σοβαρές. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή. Για να το πετύχουμε απαιτείται η στήριξη εκ των έσω προστατεύοντας αυτούς που κάνουν τις καταγγελίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζάνη. Για τους μη εγγεγραμμένους επίσης για ένα λεπτό Μπερνάρ Μονό. Ευχαριστώ. Επίτροπε, τα θέματα της φορολογίας δείχνουν ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις απαράδεκτες όπως το LuxLeaks κτλ. Αν δεν είχαν υπάρξει οι καταγγελίες δεν θα γνωρίζαμε τίποτα. Πρέπει να προστατεύουμε λοιπόν αυτούς οι οποίοι ε, διατρέχουν τον κίνδυνο παραβιάζοντας και αγνώντας τα συμφέροντά τους ε, να κάνουν τις καταγγελίες αυτές. Και αυτό θα πρέπει να μην αφορά μόνο τα φορολογικά, αλλά και το εργασιακό δίκαιο και το περιβάλλον κτλ. Όπως επίσης και τα δίκτυα σώματεμπορίας και παράνομης μετανάστευσης δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε εμείς ε, μια μαζική ε, διαδικασία κατάδοσης. Θα πρέπει όμως ε, να καταπολεμήσουμε τους απατεώνες προστατεύοντας αυτούς οι οποίοι κάνουν τις καταγγελίες. Στα πλαίσια της οδηγίας επίσης για το επαγγελματικό απόρριτο θα πρέπει να ορίσουμε σωστά τα διάφορα πεδία. Πρέπει να πετύχουμε μια ισορροπία. Η ισορροπία αυτή αν επιτευχθεί και προστατεύει και αυτούς που δίνουν τις πληροφορίες και τους δημοσιογράφους θα την υπερψηφίσουμε. Ο κύριος Ράντεφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δημιουργία μιας ιστοσελίδας στην οποία μπορούν να γίνονται καταγγελίες ε, προς την Επιτροπή την Ειδική για τα Tax Rollings είναι μια θα έλεγα επικίνδυνη πρωτοβουλία η οποία φοβάμαι ότι δεν θα δώσει τα απαιτούμενα αποτελέσματα και αυτό για διάφορους λόγους. Καταρχάς ε, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουν καταχρήσεις και να ξεκαθαρίζονται λογαριασμοί θα έλεγα μέσω των ανώνυμων καταγγελιών και νομίζω ότι τίθεται και θέμα αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει και αρνητική άποψη της ε, νομικής υπηρεσίας. Δεν θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ανωνυμία αυτών που κάνουν την καταγγελία γιατί δεν ε, έχουμε εμείς σαν βουλευτές τη νομική προστασία που έχουν δημοσιογράφοι. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα επικίνδυνο προηγούμενο το οποίο θα μπορούσε να ισχύσει και για άλλες νομοθετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές. Λοιπόν, ε, έχω την εντύπωση ότι η άποψη της νομικής υπηρεσίας είναι σωστή. Δεν πρέπει να έχουμε μια τέτοια σελίδα καταγγελιών. λεπτό η κυρία ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες δεν προστατεύουν τους ε, καταγγέλλοντες και πληροφοριοδότες. Γι' αυτό ακριβώς είχαμε τη σχετική επιτροπή για την ε, φορολογία όπου ζητήσαμε από την Κομισιόν να προστατεύσει τους πληροφοριοδότες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε επίπεδο εθνικό και διασυνοριακό και σε περιπτώσεις όπως της LuxLeaks. Είναι απογοητευτικό ένα από τα ιδρυτικά κράτη-μέλη της Ένωσης να φέρνει στο εδόλιο δημοσιογράφους ε, επειδή αποκάλυψαν αυτά τα οποία συνέβαιναν επί σειρά ετών στην ε, φορολογική διοίκηση του Λουξεμβούργου σε συνεργασία με τις εταιρείες και να μην επιτρέπεται να αποκαλύψουν πράγματα δημοσιογράφοι για... προς το δημόσιο συμφέρον. Οι αποκαλύψεις του δημοσιογράφου αυτού ήταν προς το δημόσιο συμφέρον και βεβαίως ε, πιο σημαντικές από τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας. Θα πρέπει άρα να δούμε την πρόταση Κομισιόν για ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει λοιπόν και το Λουξεμβούργο να επιδείξει λίγη κοινή λογική και να μην κατηγορεί πλέον τον δημοσιογράφο αυτό. Συγχαρητήρια στο τσακ. Λοιπόν, Μαρίζα Ματίας, τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάνουμε τη συζήτηση αυτή για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ο κύριος Περά, ο δημοσιογράφος, ε, έδωσε πάρα πολλά στοιχεία για το σκάνδαλο LuxLeaks και κατηγορήθηκε γι' αυτό. Οι πληροφορίες τις οποίες έδωσε είχαν τέτοιο βάρος που δημιουργήσαμε ειδική επιτροπή για να ρίξουμε φως στην υπόθεση αυτή. Αυτό δείχνει ε, ε, την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αυτός που θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος, είναι, θα έπρεπε να είναι ο κύριος Γιούνκερ, όχι ο δημοσιογράφος που έκανε την καταγγελία, ο οποίος θέλει να αποτρέψει ε, ε, την ε, βλάβη εις βάρος των πολιτών. Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα δεν κάνει τίποτα. Δεν προτείνει τίποτα για την προστασία των ανθρώπων αυτών. Οπότε οι πολίτες ε, θα πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα συγκεκριμένα πρόσωπα που προβαίνουν στις καταγγελίες τώρα. Σον Κέλλη. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι καταγγέλλοντες, οι πληροφοριοδότες, στα αγγλικά η λέξη προέρχεται από αυτούς οι οποίοι έχουν την ε, σφυρίχτρα, τους διαιτητές δηλαδή, ε, οι οποίοι βεβαίως δεν είναι ποτέ αγαπητοί αλλά είναι πάντοτε σεβαστοί και απαραίτητοι. Δεν είναι εύκολο και χρειάζεται θάρρος ειδικά για να αποκαλύψει κανείς ε, τέτοιες περιπτώσεις φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και μάλιστα κάποιες μεγάλες πολυεθνικές έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανές. Μιλάμε για ένα 3 εκατομμύριο το ποσό το οποίο υπολογίζεται ότι χάνεται από παράνομες μεθόδους κάθε χρόνο. Και άρα να προστατεύσουμε τους πληροφοριοδότες για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε σε δικασία και Ο Νότης Μαριάς για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή ήταν ιδιαίτερα φιδωλή στη δήλωσή της. Καταλαβαίνουμε για ποιους λόγους. Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή είναι αντικοινωνικές δράσεις και γι' αυτό πρέπει να τιμωρούνται σκληρά. Και μπορούν να αποκαλυφθούν και με τη δημοσιογραφική έρευνα αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ του δημοσίου συμφέροντος και της δημοσιογραφικής έρευνας που αποκαλύπτει τη φοροδιαφυγή διότι αυτό είναι το δημόσιο συμφέρον. η δίωξη κατά του δημοσιογράφου Εντουάν περέν είναι παράνομη είναι απαράδεκτη διότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος αποκάλυψε το σκάνδαλο των luxleaks αποκάλυψε τις ευθύνες που έχουν συγκεκριμένες χώρες φορολογική παράδειση που δίνουν την ευκαιρία στις πολυεθνικές να φοροδιαφεύγουν. επομένως η δίωξή του αυτή είναι απαράδεκτη είναι παράνομη είναι αντίθετη με την ίδια την σύμβαση την ευρωπαϊκή για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταγγέλουμε, λοιπόν αυτά τα οποία συμβαίνουν διότι αποτελούν φήμωση του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό Μιγγέλ Μιγκάς. Η φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή βρίσκονται στην καρδιά της πολιτικής και της προσοχής των μέσων ενημέρωσης. Αλλά το επίπεδο που επιτρέπει την χορήγηση πληροφοριών για ένα σάπιο σύστημα πρέπει να την χάνει κάποιας προστασίας και το δικαστικό σύστημα φαίνεται ότι έχει διαβρωθεί από τα συστήματα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής για την εξυπηρέτηση χρηματοοικονομικών συμφερόντων. Φαίνεται ότι τα συμφέροντα αυτά έχουν κυριαρχήσει έναντι όλων. Όποιος δώσει τέτοιες πληροφορίες μπορεί να φιλοκιστεί μέχρι και 20 χρόνια και να έχει πρόστιμο που να αντιστοιχεί σε μισθό χιλίων ετών. Σας ευχαριστώ. Δεν έχει δηλώσει κάποιος άλλος να ότι θέλει τον λόγο, οπότε δίνω ξανά το λόγο στην Κομισιόν. Κυρία Γιώργα. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι για τη συζήτηση αυτή. Δεν θα ήθελα να δοθεί εντύπωση ότι η Κομισιόν δεν κάνει τίποτα. Σας είπα ότι έχουμε πολλά νομοθετήματα για την προστασία των πληροφοριοδοτών που συμπεριλαμβάνουν και αυτό το θέμα. Αυτά που ακούστηκαν εδώ ότι πρέπει να γίνουν σεβαστοί οι πληροφοριοδότες διότι παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την κοινωνία, για την ένωμη τάξη κλπ ότι πρέπει να προστατευθούν δηλαδή. Συμφωνώ και είπα πριν ότι πρέπει να γίνει προστασία αυτή μέσω της νομοθεσίας. Όσο για το ευρωπαϊκό επίπεδο σας έχω ήδη πει ότι η προστασία συμπεριλαμβάνεται στην οδηγία για την κατάχρηση των αγορών και εκεί αναφέρεται και το θέμα της προστασίας δεδομένων προσωπικών ημίν Έχουν δοθεί και οδηγίες στα κράτη-μέλη για την προστασία των πληροφοριοδοτών μέσα στα πλαίσια της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων. Και η οδηγία για το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος που ενεκρίθη τον περασμένο Δεκέμβριο μιλάει και εκείνη για τους πληροφοριοδότες που τους θεωρούμε πολύ σημαντικούς. Για το Λουξ τώρα που αναφέρατε πολλές φορές, ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι η Κομισιόν δεν μπορεί να παραέμβει σε συνομοθεσία των χωρών μελών The case of, uh, uh, which... και παρόλα αυτά Έχουμε αναλάβει, έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αυξηθεί η διαφάνεια για τα φορολογικά, για την πρόληψη, δηλαδή την πρόληψη, για να καταπολεμηθεί η φοροαπαλλαγή και φοροδιαφυγή. Όσο για την προστασία των πληροφοριδιωτών σε ενωσιακό επίπεδο, θέλουμε να ληφθούν τέτοια μέτρα ώστε το κοινό να μπορεί να παίρνει τις πληροφορίες με πολύ διαφανή τρόπο. Επίσης, ήδη λάβαμε το πρώτο μέτρο που αφορά την ε, χορήγηση των πληροφοριών από τα κράτη-μέλη στην Κομισιόν για να καταχωρηθούν σε κάποιο μητρό, κεντρικό μητρό, έτσι ώστε να ξέρουμε ποια φορολογικά μέτρα έχουν ληφθεί. Και ως δεύτερο βήμα η αναχώρα αναφορές και εκθέσεις και εκ μέρους των εταιριών τα στοιχεία θα, που θα αξιολογούμε, θα αξιολογήσουμε τους επόμενους μήνες για να είμαστε βέβαιοι ότι τα μέτρα θα επιτυγχάνουν όντως το στόχο τους, δηλαδή την διαφάνεια και την πλήρη πληροφόρηση για τους Ευρωπαίους παλίτες. Αυτά τα πρώτα αποτρεπτικά βήματα ελπίζουμε να μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή και βέβαια και την προστασία των πληροφοριοδοτών και αυτό και αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.